Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα μπει στα πρακτικά τη συνεδρίαση ε, αυτό ο διορισμό. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, εγκρίνεται ο διορισμό.